οι παρεμβάσει των αντιπρόεδρων Σεύκοβιτ και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα αυτό στην Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Ελπίζω οι επισκέπτε να κατάλαβαν όλοι ότι περιμένουμε αν θέλουν να καταθέσουν πρωτοβουλίες ε, σε συνεργασία με πολίτες 7 χωρών. Ε, Μην διστάσετε λοιπόν, ε, περιμένουμε τις πρωτοβουλίες. Ανακοίνωση. Το ΕΛΚ ζητεί ο κύριος Φαμπρίτσιο Μέρτον να οριστεί μέλος της Επιτροπής ε, ε, Βιομηχανίας Έρευνας Ενέργειας. Παρατηρήσεις όχι. Εγκρίνεται λοιπόν αυτός ο διορισμός του. Και ακολουθεί τώρα η συζήτηση της προφορικής ερώτησης ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Καταφθάνει η κυρία Μπόλς Περιμένουμε λίγα λεπτά, γιατί είναι εκείνη η συντάκτρια της ερώτησης και οπότε είναι δύσκολο να αρχίσουμε απουσία της. À votre aise, Madame Bose, ne tombez Είστε συντάκτρια της ερώτησης και θα πάρετε το λόγο ως εκ τούτου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι ο Επίτροπος ε, δεν μπορεί να είναι στη διάθεσή μας διότι μεταβαίνει τώρα στην Ουάσιγκτον. Ε, φαίνεται όμως ότι επαναλαμβάνονται αυτά τα φαινόμενα ότι δεν μπορούμε ενώπιον ε, του Επιτρόπου να κάνουμε τη συζήτησή μας γιατί πάντοτε πέφτει την Πέμπτη και πάντοτε κάπου είναι. Λοιπόν, με την ε, δέσμη έξι οδηγιών ε, θεσπίσαμε το σύστημα αντιμετώπιση των μακροοικονομικών δυσκολιών για να εφαρμοστεί σωστά το σύμφωνο σταθερότητα. Η επιτήρηση ήδη επεκτείνεται στα μακροοικονομικά ζητήματα πέραν του ελλείμματο δηλαδή και του χρέου όπω ίσχυε μέχρι τούδε. Και έχουμε και τον πίνακα επιδόσεων με δείκτε που λειτουργούν ω διαγνωστικό σημαντικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Νοέμβριο του 2012 στο αρχικό σετ προδιαγραφών προσετέθη ένας νέος δείκτης για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και για την αστική ευθύνη αυτού του τομέα. Now, in order to... Για να αποφύγουμε τις ε, παρανοήσεις ε, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει δείκτης, ε, ότι είναι ευπρόσδεκτος ένας τέτοιος νέος δείκτης. Το ζήτησε το Σεπτέμβριο του 2011 το Κοινοβούλιο ούτως ή άλλως. Ε, ο επιλεχθής δείκτης ε, δεν είναι πλημελής, ε, δεν ισχυρίζομαι αυτό, όμως υπάρχουν πάρα πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις και πολλοί άλλοι δείκτες. Δυστυχώς δεν τήρησε την δέσμη 6 οδηγιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εκεί υπάρχει συνεννόηση ότι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχόλια προς τις συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου και τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου για τον προγραμματισμό και θέσπιση όχι μόνο των δικτών αλλά και των κατοφλίων. Ε, σε αυτή την περίπτωση είναι ξεκάθαρο δεν έλαβε χώρα η προβλεπόμενη διαβούλευση. Το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε για το νέο δίκτυ ημέρες ε, μετά την δημοσίευσή του και ουχή νωρίτερα όταν ε, το Νοέμβριο του 2012 συστάθηκε ο μηχανισμός έγκυρης προειδοποίησης. Μα έπληξε αυτό πέρα από τον κόλαφο που συνιστά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Οικονομικής Επιτροπής πέρασε τον δικτύ χωρίς καμία διαβούλευση επιτροπές και οι υπηρεσίες τους ε, δεν μπόρεσαν ε, να τοποθετηθούν και δεν εκατοχυρώνονται τα ίσα δικαιώματα Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διαβούλευση, μας είπαν με το Κοινοβούλιο αλλά θα μπορούσαμε ε, ατύπως ε, να έχουμε λάβει το σχέδιο μέσω της Γραμματείας. Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου απέδειξε στο παρελθόν ότι είμαστε αποτελεσματικοί και συνεργαζόμαστε καλή την πίστη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ε, Προσπάθησα να διαλευκάνω το ζήτημα μέσα από ανταλλογή επιστολών μετά τη δημοσίευση του δείκτη κατά το μήνα Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Λογική εξήγηση δεν έλαβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να παραδεχτεί το λάθος της και να υποσχεθεί να τα καταφέρει καλύτερα την επόμενη φορά. Ε, διότι με τη γάμα δέλτα μάρκτη ε, ο Επίτροπος ε, Μπαρνιέ αυτό ακριβώς έκανε ε, και ε, ε, έδρασε όπως άρμοζε. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν καθόλου και τυπικά εντάξει και αυτό δεν ισχύει και εξού και η προφορική μου ερώτηση. Θα θέλαμε μία ξεκάθαρη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν διαβουλεύτηκε με το Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν προσέθεσε αυτό το δίκτυο για την σταθερότητα και τις μικροοικονομικές ανισορροπίες. Προτού προσπαθεί ο μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση το 2013 και θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το ψήφισμα τη 15 η Δεκεμβρίου του 2012 για τον πίνακα επιδόσεων για ενισορροπίε μακροοικονομικές ε, ε, δεν επαρκεί ω θέση του Κοινοβουλίου διότι εκεί προτείναμε να προσθεθεί ο χρηματοπιστωτικό τομέα και εκεί προβλεπόταν η διαβούλευση όπω προβλέπεται και από την αιτιολογική σκέψη υπαριθμών 12 ε, της διαδικασίας περί μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κυρία Μπαούλη. Απάντησε από την Επίτροπο Μάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη. Είναι λυπηρό που ο αντιπρόεδρος Ρεν ε, κολλιέται και δεν είναι σήμερα εδώ έχει ανηλυμένες χρεώσει στην Ουάσιγκτον ε, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το G20 ήταν στη διάρκεια της εβδομάδας εδώ όπως γνωρίζετε αλλά υποχρεώθηκε να φύγει. Σε σχέση με την ερώτησή σας, όπως είπε η αξιότιμη βουλευτής ε, ε, αυτό ήταν αντικείμενο αλληλογραφίας που είχατε με τον αρμόδιο επίτροπο 4 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία, δεν θα επαναλάβω τα όσα λέγει η επιστολή, τα γνωρίζουν όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ε, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λυπάται για την ε, θεώρηση που έχει το Κοινοβούλιο ότι ε, δεν διαβουλεύθηκε μαζί του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ε, δεν ήταν η πρόθεσή μας, ούτε αντιλαμβανόμαστε έτσι ε, την ε, εξαγωγή αυτή. Ε, επιλέξαμε τον 11ο δίκτυ ε, σύμφωνα με την πολιτική συμφωνία που είχε ήδη επιτευχθεί τέλη του 2011 με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τη συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων. Θυμίζω ότι με βάση αυτόν τον κανονισμό είναι ρόλος και καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσαρμόζει ε, τον ορισμό του πίνακα επιδόσεων. Και παραθέτω όταν χρειάζεται μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οφείλει να αλλάζει τη μεθοδολογία, τους δείκτες να προσαρμόζει ή να τροποποιεί ε, όταν αυτό και όπου χρειάζεται. Τέλος της παράθεσης. Στενή συνεργασία με το Συμβούλιο ε, και με το Κοινοβούλιο είναι το πνεύμα που διέπτυσε συνεργασία μας και εκ των όνου το αναφέρει και η ιδεολογική σκέψη 12α. Ε, είστε δύο συνομοθέτε για τα χρηματοπιστωτικά και το 2011 επετέφθη συμφωνία μέσω ψηφίσματο του Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου και ε, των συμπερασμάτων του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ το Νοέμβριο του 2011. Τονίζω αυτή τη σημασία. Οι πολιτικέ επιλογέ έγιναν το 2011 από κοινού με το Κοινοβούλιο. Το 2012 ήρθε η ε, τεχνική υλοποίηση. Προσετέθη ένα δείκτη χρηματοπιστωτικού τομέα στον πίνακα επιδόσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί ότι θεωρεί ότι η διαβούλευση έγινε το 2011 και ότι το τότε ψήφισμα του Κοινοβουλίου ήταν η πολιτική απάντηση στα διακυβευόμενα. Έχουμε ίση μεταχείριση και προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, τους ενημερώνουμε ταυτόχρονα και ε, λαμβάνουμε υπόψη ε, όσα λέγει η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, η PC η οποία είναι συμβουλευτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλο εξ τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να πω σε όλους τους βουλευτές ότι έχουμε αναλογική ε, προσέγγιση. Χώρες αντιμετωπίζουμε διαφορετικό τρόπο μακροοικονομικές ισορροπίες. Ε, ο πίνακας επιδόσεων θα πρέπει ε, να είναι καλά σχεδιασμένο και να εφαρμόζεται σωστά. Ε, άνθρωποι είμαστε, κάνουμε σφάλματα. Ε, δεν υπάρχει κανένας δείκτης που να ε, μπορεί να μετράει από μόνος του τις δυσκολίες του χρηματοπιστωτικού τομέα και τι επιπτώσει στην πραγματική οικονομία. Γι' αυτό δεν είναι ποτέ μηχανικός ή αυτόματος ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τον πίνακα επιδόσεων. Υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο δικτών που αναπροσαρμόζονται, που ε, χρησιμοποιούνται και όπως γνωρίζετε δημοσιεύτηκε στις 10 Απριλίου. Ελπίζω αυτά που σας είπα να ε, διευκρινίζουν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόρφμαν έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, αξιότιμη συνάδελφοι κυρίες και κύριοι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το 2011 εγκρίναμε τη μακροοικονομική εποπτεία. Στο μεταξύ εφαρμόζεται το εργαλείο αυτό και είναι πάρα πολύ κομβικό μέσο της κοινή οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον. Το 2011 είχα την τιμή να συμμετέχω στην εκπόνηση του κανονισμού και ήδη από τότε το πάρα πολύ βασικό θέμα ήταν ποιο ρόλο διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εκπόνηση του πίνακα επιδόσεων, scoreboard, η βαθμολόγιο. Και λυπάμαι πάρα πολύ που απουσιάζει ο κύριος ε, Ρεν, γιατί είχε δεσμευτεί τότε και μόνο βάσει αυτής της δέσμευσης το Κοινοβούλιο έδωσε τις ευλογίες του για τον κανονισμό. Ήμασταν υπέρ μιας ε, ευέλικτης ε, μορφής χειρισμού με σχέση εμπιστοσύνης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά στις 19 10 κοινοποιείται στο Κοινοβούλιο ότι έχετε προσθέσει νέο δίκτυ και μετά από μία εβδομάδα θα αρχίσετε να το χρησιμοποιούτε. Δηλαδή, ε, το ξέρατε μήνες χωρίς να ενημερώσει το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι χοντρό φάουλ περί τίνος πρόκειται. Εδώ είμαι στο πλευρό της συναδέλφου Προέδρου της Επιτροπής μας, κυρίας Μπόουλς. Το θέμα δεν είναι ο δείκτης αυτός καθ' αυτός. Δεν θέλουμε κοινοβουλευτική συζήτηση κάθε φορά, αν θα προσθετήθεται ένας δείκτης. Ε, ούτε θέλουμε νέους δείκτες. Γι' αυτό έχουμε κάνει ε, την πρόταση να μην υπερψηφίσουμε την τροπολογία αυτή. Άρα, τι μας ενδιαφέρει εμάς. Ε, για να το πω ε, έτσι κάπως χοντρά, δεν θέλουμε να παρουσιάσουμε την παρεξηγημένη παρθένα, αλλά θέλουμε να συμμετέχουμε στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, θα πρέπει να έχουμε αποδοχή στα μάτια των πολιτών. Αποδοχή στα μάτια των πολιτών δεν υπάρχει χωρίς δημοκρατική εξασφάλιση. Αυτό είναι το θέμα. Και σας το λέγω γιατί εγώ προέρχομαι από μια χώρα που είναι η Ιταλία και αυτό το θέμα της αποδοχής και της εμπιστοσύνης στα μάτια των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος θέλει να έχει την αίσθηση ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ ε, είναι καλυμμένε κοινοβουλευτικά και εξασφαλισμένε ότι έχει προηγηθεί δηλαδή η κοινοβουλευτική συζήτηση. Και τώρα εσεί τι ζητάτε από εμά, να βγούμε εμεί οι βουλευτέ τώρα προ τα έξω, στα κράτη-μέλη και να πούμε ότι υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία. Ε, δεν μπορούμε να το πράξουμε αυτό. Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διονύζει αυτή την εικόνα ότι την Ευρώπη την κυβερνάει η γραφειοκρατία. Και είναι κρίμα. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη στιγμή που ε, ε, καλούμαστε να εξηγιάνουμε την οικονομία μας και είναι δύσκολη η κατάσταση, χρειαζόμαστε νέα αφετηρία. Με αυτή τη διαδικασία και την τακτική σίγουρα δεν το εξασφαλίζουμε αυτό. Εμείς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά πιστεύω και το Κοινοβούλιο συνολικά, επιθυμεί να επιτύχει η μακροοικονομική εποπτεία. Εσείς με αυτή τη συμπεριφορά και την τακτική σίγουρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχετε συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε τα εξή από το Κοινοβούλιο. Τα εξή τέσσερα. Διαφύλαξη πρώτον του ρόλου του Κοινοβουλίου. Σιγά σιγά θα πρέπει να το αντιληφθεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε, έχουμε μια συνθήκη που λέγεται τη Λισαβόνα. Ε, δεύτερον, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι όργανα ισότιμα και θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Δεν έγινε εδώ. Τρίτον, ποιος είναι ο ρόλος του ευρωπαϊκού συστήματος ε, συστημικού κινδύνου. Δεν έχει ληφθεί υπόψη σοβαρά και τέταρτον, σε κάθε μελλοντική προσαρμογή, που ε, αναφίβολα θα υπάρξει, γιατί αυτό που αναφέρατε για ε, την ευελιξία και των δικτών και του πίνακα επιδόσεων, κυρία Επίτροπε, είναι σωστό οποιαδήποτε περαιτέρω προσαρμογή θα πρέπει να ανακοινώνεται εγκαίρως όμως το Κοινοβούλιο για να έχουμε ε, αποτελεσματική συζήτηση όπως είπε και η Πρόεδρος Μπόλτς. Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση. Φροντίστε αυτά που ζητούμε να λειτουργούν αποτελεσματικά και να στεφθούν με επιτυχία όλες αυτές οι διαδικασίες για την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Ντόρφμαν. Η κυρία Φερέιρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε. Το πρόβλημα που τίθεται εδώ είναι ένα πρόβλημα ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη από πλευρά των δύο θεσμικών οργάνων για τι νομοπαρασκευαστικέ διαδικασίε. Ε, η συγγήτρια για αυτό ακριβώς το θέμα, για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν τεχνικά και πολιτικά ζητήματα. Είναι δύο διακριτές ε, ομάδες. Η επιλογή των δικτών και των κατοφλίων για την έγκαιρη προειδοποίηση είναι ένα πολύ ε, τεχνικό ζήτημα. Επί τη βάση αυτών των πληροφοριών ε, καταρτίζονται οι πολιτικές ή τροποποιούνται αυτές οι πολιτικές. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή επιλογή των δικτών είναι μία απόφαση εξαιρετικά σημαντική για να γνωρίζουμε βάσει των αποτελεσμάτων, βάσει αυτών που έχουμε συμφωνήσει, να μπορέσουμε να λάβουμε τις δέουσες αποφάσεις. Ε, ε, Επίτροπε, Αναφερθήκατε σε αυτό το έγγραφο, στην αιτιολογική σκέψη υπαριθμών 12 και θα σας το διαβάσω στα αγγλικά, λέει η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει προτάσεις προς σχολιασμό στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με στόχο τη θέσπιση και προσαρμογή δικτών και αριθμητικών κατοφλίων. Συνεχίζω στα πορτογαλικά. Γι' αυτό και... Ε, ε, αυτό είναι στη βάση της διαθεσμικής μας ε, συμφωνίας ε, και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί δεν είχαμε ενημέρωση για την προσαρμογή του δίκτυ. Επίτροπε, θεωρείτε ότι έτσι τηρείται το πνεύμα και το γράμμα της λόγω αιτιολογικής σκέψης. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρεί τον τρόμο με τον οποίο ερμήνευσε αυτή την προσαρμογή και ότι θα επανορθώσει το σαφές σφάλμα που διέπραξε βάσει βάση της διοργανικής συμφωνίας, διότι εγώ θεωρώ ότι διεπράχθη τέτοιο σφάλμα και οφείλει να το αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα προσθέσω περισσότερα. Νομίζω ότι η, Επιτροπή ε, η, συγγνώμη, η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, η κυρία Μπόλς, το εξήγησε αρκούντος. Ε, θεωρώ ότι θα χρειαστούμε μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο συνεργασίας των θεσμικών οργάνων διαφορετικές φάσεις γιατί είναι πολυάριθμες είναι απολύτως απαραίτητο να μετάσχουμε επί τη βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρο. Σας ευχαριστούμε κυρία Φερέιρε, η κυρία Σιλβί Γκουλάγ από πλευράς των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που είσαστε εσείς σήμερα ως πρόεδρος. Για ποιο λόγο η ε, κυρία Επίτροπος, για, για ποιο λόγο, για τη λογικότητα της Κομισιόν και το θέμα που συζητάμε σήμερα, όπως είπε η Λίζα και άλλοι προηγουμένως, είναι η ίδια η φύση των σχέσεών μας. Σε αυτή λοιπόν την Ευρώπη, όπως είναι αυτή τη στιγμή με τι συνθήκε τη κλπ. κλπ αποδεχόμαστε το ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε ή όχι. Περί αυτού πρόκειται. Δεν νομίζω να είναι περίπλοκο το θέμα, δεν είναι τεχνικό ή τεχνοκρατικό. Υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμού, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα χωρίς να περιπλέκουμε τα πράγματα. Και εγώ ήμουν εισηγήτρια για την εξάδα των μέτρων και θα μπορώ να σας πω ότι είχαμε μια μακροχρόνια διαπραγμάτευση και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η διαδικασία αυτή να διεξάγεται υπό καλό πνεύμα συνεργασίας. Μπορέσαμε να καταθέσουμε κείμενα μεταξύ των τριών. Γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τους δείκτες και να τους οριστικοποιήσουμε. Εδώ έχει ένα θέμα, έχουμε ένα θέμα ουσίας. Ποιο είναι το διακύβευμα. Δεν ε, έχουμε να κάνουμε ας με ελοξυπηρετήσεις. Μέχρι τώρα στην ε, ζωή του ευρώ όλοι αποφασίσαμε να έχουμε μία προσέγγιση η οποία όμως μέχρι τώρα ήταν περιοριστική που κοίταζε περισσότερο το χρέος. Με την εξάδα των μέτρων για πρώτη φορά έχουμε εργαλεία ώστε να κάνουμε εξοικονομήσει μαζί. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν από κοινού τι λειτουργεί και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο και επιπτώσει στην ζωή των πολιτών. Δηλαδή υπάρχει ας πούμε ανεργία, το επίπεδο εισοδημάτων, μισθών των εργαζομένων είναι δίκαιο Αυτά είναι τα θέματα που καίνε του πολίτε. Αν λοιπόν το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση τουλάχιστον να μεταφέρει αυτά τα αιτήματα ή να στείλει μηνύματα, τότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω ποια άποψη θα υπερισχύσει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα, ένας χώρος συζήτησης, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό θα τελειώσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και βλέπουμε να υπάρχει μια αύξηση της αμοιβαίας της πιστίας είτε πρόκειται για ε, αισθήματα που προχωρούν από το Βερολίνο είτε από τις Βρυξέλλες δημιουργεί έτσι μια αμοιβαία πικρία. Ή λοιπόν από κοινού θα δράσουμε μαζί και θα ε, υιοθετήσουμε τα απαραίτητα να το κάνουμε αυτό, διαφορετικά θα πέσουμε πάνω στον τοίχο και θα καταστραφούμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά θέματα ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, οικονομία και όχι μόνο θέματα αμοιβαίου ελέγχου όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φιλίπ Λαμπέρξ, ονόματο των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Άννη. Ε, θα μπορούσα να προσυπογράψω όλα όσα είπε τώρα η Σιλβή. Κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, σε εσά απευθύνομαι. Κυρία Επίτροπε, άκουσα τα ωραία σα λόγια και ο ίδιος ο συνάδελφός σας ο Λιρέν τα ίδια ωραία μα λέει. Δεν σας πιστεύω ούτε λέξη. Ε, όταν εγκρέατε το πρώτο βαθμολόγιο πάλι μας, περιπέξατε, μας περιγελάτσατε το ίδιο κάνετε και τώρα το είχαμε πει ε, δεχτήκαμε να απεμπολίσουμε την συναπόφαση ε, σε αυτό το θέμα από εμπιστοσύνη και την προδώσατε αυτή την εμπιστοσύνη δις παρακαλώ σήμερα η εμπιστοσύνη που έχουμε σε εσά είναι μηδενική και μένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην βάζει στο δίκτυο επιδόσεων βασικά θέματα. Το μόνο που του ενδιαφέρει στην παραγωγικότητα είναι η παραγωγικότητα τη εργασία. Ξεχνούν την παραγωγικότητα των πόρων, τη ενέργεια και όλου τυχαίω και την παραγωγικότητα του κεφαλαίου. Και όλου τυχαίω επίση τι ανισότητε να μην τι δούμε ε, 25% στην Ευρώπη των ανθρώπων ζουν ε, κάτω από το όριο της φτώχειας. Και εσείς ε, κοιτάτε αλλού. Η Ευρωπαϊκή πρέπει να αλλάξει και γνώμη, αλλά θα πρέπει να αλλάξει και το βλέμμα με το οποίο βλέπει τα πράγματα. Καθόμαστε πάνω σε μια βόμβα. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω και πολλοί άλλοι στο Κοινοβούλιο, έχω σοβαρότατε ανησυχίε σε σχέση με τη μεταχείριση που μα επιφυλάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίω για αυτό το ζήτημα, αλλά όχι μόνο. Για κάποια ζητήματα, όπω παραδείγματο χάρη μεταρρύθμιση νομοθεσία ε, για τα παράγωγα. Ε, πρόκειται για τη νομοθεσία επίπεδου 1, αλλά αυτό προποθέτει ότι θα ληφθούν και αποφάσει για το επίπεδο 2 και δεν μπορεί να παρακάμπτεται το Κοινοβούλιο υιοθετώντα ε, αποφάσει ε, τόσο σύντομα σύντομα, ώστε να μην έχουμε εμεί χρόνο για να τι ε, σχολιάσουμε. Και αφήστε, δεν μιλάμε καν για ουσιαστική διαβούλευση και σχολιασμό το Κοινοβούλιο. Πράξη κατά σε εκτελεστικά μέτρα, τεχνικέ, ε, τεχνικά εφαρμοστικά μέτρα. Καταλαβαίνετε, οι πολίτε στην εκλογική μου περιφέρεια ούτε που ξέρουν τι ακριβώ σημαίνουν αυτά τα πράγματα. 98% τη ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, έτσι παράγεται αυτή τη στιγμή και βάσει αυτών των εκτιμήσεων, 10 άτομα εδώ στο Κοινοβούλιο και 50 εκτό Βρυξελών κατανοούν ε, το πώ λειτουργεί το σύστημα. Καταλαβαίνετε ε, γιατί μα κατηγορούν ότι δεν είναι δημοκρατικό ο τρόπο ε, και η διαδικασία λήψη αποφάσεων. Μα αυτός δεν είναι ο στόχο. Ο στόχο είναι να είναι πιο ευέλικτη η νομοθεσία και να προσαρμόζεται σε όλε τι αλλαγέ θεωρητικά. Συμφωνώ με αυτό και υποστηρίζω την αρχή. όμω, αν αυτό δεν συμβεί με ένα γνήσια δημοκρατικό τρόπο τηρώντα το πνεύμα τη συνθήκη, αλλά και το γράμμα τη. Ε, πρόκειται για ε, ε, επιταγές που μεταφράζονται σε νομοθεσίες σε διαταγές που μεταφράζονται σε νομοθεσίες. Αυτό συνέβη στην περίπτωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και του ε, πίνακα επιδόσεων. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ε, μετρήσεως ε, και οι τρόποι υπολογισμού, παραδείγματο χάρη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν ταυτίζονται με τον τρόπο υπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταλαβαίνετε ότι αυτό καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σοφότερη όλων. Στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη εμπιστοσύνη του ε, και αυτός δεν είναι ο σωστός δρόμος. Χρειάζονται ορθότερες διαδικασίες ε, ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στους συνομοθέτες και να εξασφαλίζεται ένας ε, δημοκρατικός έλεγχος σε αυτήν την διαδικασία. Σας ευχαριστούμε κυρία Σουίνμπουρν, δεν βλέπω τον κύριο Κλούτε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ζάλιστρα από τους μη εγγεγραμμένου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο είναι οργισμένο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην προσαρμογή του πίνακα επιδόσεων μετά τη δέσμη έξι ε, ε, οδηγιών. Χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κράτη-μέλη και το Συμβούλιο ε, για να δουν αν τηρούνται τα υποσχεθέντα. Όταν εγκρίθηκε το Six Pack, ε, ε, το κόμμα μου ήταν κατά, γιατί περιστέλλεται η εθνική κυριαρχία. Η εθνική κυριαρχία είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, όχι να το απεμπολούμε. Ε, αυξάνεται η ανεργία, μειώνεται το έλλειμμα. Δεν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μετράει τέτοιους δείκτες. Τι νόημα έχει ο δείκτης επιδόσεων για να δείχνουμε ότι η Ευρωζώνη δεν είναι σταθερή. Ε, κυριαρχεί η Γερμανία, αλλά δεν φταίει η Γερμανία που οι άλλε χώρε δεν είναι ανταγωνιστικές. Είναι χώρε που δεν μπορούν να κάνουν την οικονομία του ανταγωνιστική. Δεν βοηθούνται από ένα δίκτυ ή από ένα πίνακα επιδόσεων. Ε, στην Ευρωζώνη δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Αν δεν μπορούν να φύγουν. Και αυτό είναι προς το καλό και της χώρας και των πολιτών. Αυτό που μας ενδιαφέρει ε, είναι η ε, διαδικασία ε, και δεν συζητούμε τι σημαίνει η εκχώρηση αρμοδιοτήτων προς τις Βρυξέλλες. Δυστυχώς ε, αυξάνεται η εκχώρηση αυτής της κυριαρχίας. Η διαδικασία δεν έχει νόημα. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καταλάβουν ότι είναι δική τους ευθύνη η θέση τους στον κόσμο και η ευημερία των πολιτών τους. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στου υπόλοιπου εγγεγραμμένου ομιλητέ. Πρώτα θέλω να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Γκουαλτιέρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η υπόθεση με την ε, έλλειψη διαβούλευση στο Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτούς τους ε, δείκτες δεν είναι σοβαρή από μόνη της, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα γενικότερο μήνυμα του λανθασμένου τρόπου με τον οποίο η Κομισιόν αντιλαμβάνεται τον δικό της ρόλο και την ε, σχέση με το Κοινοβούλιο υπό το φως των λέων αρμοδιοτήτων όλα την χρηματοοικονομική διακυβέρνηση που ανέλαβε μετά την κρίση. Αυτό είναι το κύριο πολιτικό ζήτημα όπου το επεισόδιο αυτό αποτελεί άλλο ένα μήνυμα. Και πίσω από αυτό το επεισόδιο, πίσω από αυτή την υπόθεση, τη μεθοδολογική, υπάρχει ένα θέμα πιο βαθύ, πιο πολιτικό. Εμείς είμαστε δυσαρεστημένοι για τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν χρησιμοποιεί την διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να καταδείξει τις ανισορροπίες όσον αφορά την αλληλοεξάρτηση και την αμοιβαιότητά τους. Ε, τα θέματα του χρέους και των πλεονάσματων, το αυξανόμενο κόστος εργασίας σε σχέση με την παραγωγικότητα, αλλά και την εργασία η οποία αυξάνεται ελάχιστα. Αντίθετα, η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα του Συμφώνου Σταθερότητας βασίζεται ακόμα στην φιλοσοφία των ενάρετων και των μη ενάρετων. Και αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Γιατί χωρί μια κατάλληλη σχέση με το Κοινοβούλιο θα είναι δύσκολο να διορθώσουμε τι βαθιέ ζημιέ που θα έχουμε όσον αφορά την ποιότητα τη χρηματοοικονομική μα διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Αδελφός Κλίβα, για ένα λεπτό. Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ευχαριστώ. Θα έπρεπε να εμπλακεί αμεσότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την επιλογή των δικτών για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ε, θα συμφωνήσω λοιπόν με τους προλαλήσοντες. Ε, ο πίνακας επιδόσεων για διαδικασία ε, μακροοικονομικών ανισορροπιών θα πρέπει να είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εντελεχή ανάλυση της κατάστασης και πρέπει να συνυπολογίζεται ατυχώς ε, παρά την ανακοίνωση που προηγήθηκε για τη Σλοβενία μεταξύ άλλων δεν βλέπουμε καμία σχέση ανάμεσα στην αποτίμηση της εθνικής ε, κατάστασης αφενός και αφεντέρου τα πολιτικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως αυτά έχουν κέρια σημασία, ε, έχουν μεγαλύτερο ειδικό βάρος σε σχέση με μελέτες του ΩΣΑ, παραδείγματο χάρη. Θα έπρεπε λοιπόν να εμπλακεί άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποστηρίζω την έκκληση βάσει της οποίας ε, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας επιτήρησης των μακροοικονομικών ανισορροπιών θα πρέπει να επικρατήσει το δημοκρατικό στοιχείο και να ακούγεται η άποψη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε η πρόληψη και η διόρθωση των μακροοικονομικών ισορροπιών που είναι υπερβολικέ, νομίζω αποτελεί ένα βασικό πυλώνα τη ε, χρηματοοικονομική διακυβέρνηση τη Ευρώπη. Απαιτεί διαφάνεια και μια δημόσια διαδικασία δημοκρατικών αποφάσεων που θα προασπίσει τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να εφαρμόζεται με, το, με τη συμμετοχή και τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θέσπιση δικτών αποτελεί ένα πολιτικό εργαλείο υψίστου επίπεδου. Ένα θέμα δημοκρατικό και όχι γραφειοκρατικό γιατί με αυτόν τον τρόπο εντοπίζουμε σαν ισορροπίε, διασφαλίζουμε την σωστή λειτουργία του μηχανισμού αγκές περιτοποίηση και κάνουμε διαφορετικά μέτρα. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να τα εφαρμόσει όλα αυτά στα πλαίσια μια κοινοβουλικής δημοκρατία που ε, περιλαμβάνει και λαμβάνει υπόψη και τις ε, συνενέσεις. Τρία μηνύματα λοιπόν. Πρώτον, τα δεδομένα, μάλλον τα τα τετελεσμένα προς το Κοινοβούλιο είναι κάτι απαράδεκτο. Μετά, η έλλειψη μεταξύ ίση ίσης μεταξύ των συνο, ε, συνομοθετών και τρίτων δεν μπορούμε να αναβάλουμε ε, την ανισορροπία μεταξύ των χωρών που έχουν πλεόνασμα και χωρών που έχουν χρέο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας Catch the Eye. Ε, πρώτα θα καλέσω τον κύριο Κούτας να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που εκφράζουν επικρίσει. για το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε για την προσαρμογή του πίνακα επιδόσεων για την εποπτεία ε, σε σχέση με τα πρόσφατα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στις, 11, στις 10 Απριλίου. Ε, λυπούμε που ε, δεν κοιτούν τα πλεονάσματα στη Γερμανία, για παράδειγμα, γίνεται λόγος για 6% το ΕΠ πλεόνασμα. Δεν το συμπεριλαμβάνουν στην ανάλυση τους. Επίσης δεν κοιτούν τη σχέση ε, μεταξύ παραγωγής και κόστους παραγωγής και μισολογικού κόστους και αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να ε, συγκρίνονται. Όταν μιλούμε για ανισορροπίες μεταξύ ε, οικονομιών θα πρέπει να κοιτάμε τις χώρες περιφέρειας και τις χώρες του κέντρου και θα πρέπει να υπάρχει και αύξηση μισθών σε κάποιες χώρες. Όλα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστώ. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες ε, στη κρίση του χρέους μπορεί να έπαιξαν ρόλο, γι' αυτό και η κρίση μας έδωσε ένα οδυνηρό ε, μάθημα. Η οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία διατάσσονται ε, από διατάγματα ούτε από επιταγές της Τρόικα και καμία οικονομική διακυβέρνηση ε, δεν πρόκειται να πετύχει. Θα αποτύχει η κτρά. Είναι πολύ διαφορετικέ οι προποθέσει από χώρα σε χώρα. Δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε αυτά. γεγονό είναι ότι κάθε κράτο μέλο θα πρέπει να ανταποκρίνεται με το δικό του τρόπο στι ιδιαίτερότητε που έχει. Και έχει φτάσει η ώρα ε, να ε, αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις διαφορές της χώρες ως ενίσχυση και να μην τα ισοπεδώνουμε όλα για να είμαστε όλοι ομοιόμορφοι. Ε, και είναι από μόνο του ε, αμφισβητήσιμο το γεγονός ότι μεταφέρουμε πόρους σε χώρους που έχουν χρέη. Ε, και δείχνουμε, φαίνεται πιανού πνευματικό παιδί είναι η Ευρώπη σήμερα. Ευχαριστώ. Εξ ονόμας Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επίτροπο Μάλστρομ, ευχαριστώ αξιότιμοι βουλευτέ για τη σημερινή συζήτηση. Με, μου απευθύνατε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον για την παραγωγικότητα να ε, ενταχθεί στο πεδίο ή για τον μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση. Μα περιλαμβάνεται η παραγωγικότητα, αλλά είναι συμπληρωματικός δείκτη, όπω και άλλοι δείκτε, όπω οι επενδύσει, ε, ε, οι επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη, ε, οι μονάδες εργατικού κόστους ε, που συνυπολογίζονται στο εργατικό κόστος καθώς και παραγωγικότητα. Για τη συμμετρία που με ρωτήσατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εφαρμόζει αυτή την ευφυΐα συμμετρία όπως ονομάζεται για τα ελλείμματα, τα τρέχοντα ελλείμματα και τα τρέχοντα πλεονάσματα. Υπάρχουν όμως διαφορές διότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια πλήρη συμμετρία. Έχουμε εκπονήσει ολάκερη έκθεση για αυτό το ζήτημα και σας παραπάνω αυτήν. Uh, Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Όπως σας είπα και νωρίτερα και αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσδίδουμε ύψη τη σημασία στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και όταν κατά την επιλογή των μακροοικονομικών δικτών ουδόλως είχε την πρόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακάμψει το Κοινοβούλιο. Η προθεσμία για την κοινοποίηση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μικρή και αυτό εξηγείται στο ότι οι τεχνικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου και αφετέρου Είμαστε απολύτω πεπισμένοι, ήμασταν απολύτω πεπισμένοι ότι είχε δώσει το πράσινο φω ε, το Κοινοβούλιο ήδη. Ε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε εγκαίρω να έχουμε προετοιμάσει τον δείκτη για την δημοσίευση τη μελέτη για το μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση, όπω είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο. Ε, και δύσκολα μπορεί κανεί να ερμηνεύσει διαφορετικά τι προσπάθειε που έχουμε κάνει. Είναι καλόπιστε, ε, πιστέψτε μα, για τι μελλοντικέ τροποποιήσει του πίνακα επιδόσεων για τι μακροοικονομικέ ανισορροπίε. Θα ακολουθήσουμε ακολουθήσουμε ακριβώ την ίδια οδό, διότι συμφωνούμε απολύτω ε, ότι μόνο μέσω τη συνεργασία μπορούμε να προχωρήσουμε και όταν αμοιβαίω ενισχύουμε και την αξιοπιστία και τι αρμοδιότητε ε, των θεσμικών ε, οργάνων τη Ένωση. σε κάθε πιθανή ευκαιρία θα πρέπει με αναλογικό και επικοδομητικό τρόπο να επιδιώκουμε την διοργανική συνεργασία και όπως γνωρίζετε ο Αντιπρόεδρος Ρενέ θα έρθει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων Υποθέσεων ε, σύντομα και θα μπορέσει να συζητήσει περαιτέρω αυτό το τεχνικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε Επίτροπο Μάλμστρομ. Η συζήτηση ε, έληξε. Το Προεδρείο έχει λάβει μία πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση της συζήτησης και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30. Η συνεδρίαση διακόπτεται μέχρι την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ.